Παραλαμβάνει τη συνεδρίαση που διακόπηκε 16 Φεβρουαρίου 2010. Κυρίες και κύριοι, πριν από ένα έτος ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη, η οποία έφερε ελευθερία σε πολλούς από τους νότιους γείτονές μας και στη Συρία